say uh, in our let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de cette. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη που έχουμε αλλαγέ την τελευταία στιγμή, που αργήσαμε. Σας ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Σημείο 14. Δίνω το λόγο. Μάρτιν Κάσλερ, πού είναι? Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Μια στιγμή. Ξέρω, θα είναι η κυρία Γέγκλερ. Εντάξει, αντικαθιστάμε τον κύριο Κάσλερ. Όπως είπαμε και χτες, στην πραγματικότητα το πρώτο σημείο για σήμερα θα είναι το σημείο 13α και που έχει να κάνει με την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα και το σημείο 19 που θα ψηφίσουμε και με την εξέταση των τροπολογιών του σημείου αυτού. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων έχει αρχίσει να δουλεύει πάνω στην επαναδιατύπωση του άρθρου 81 του κανονισμού. Είναι το άρθρο το οποίο καθορίζει τις ε, προϋποθέσεις εξέτασης από το Κοινοβούλιο ε, γράφων για το οποίο δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Αν δείτε λοιπόν τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο όπου η σποδηλική στήλη στην εξέταση των κειμένων είναι τα συνήθη κείμενα, νομοθετικά ή μη, και στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες διαδικασίες οι οποίες προσαρμόζουν την νομοθετική ή μη νομοθετική διαδικασία κατά περίπτωση όπου πρέπει να αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, δημοσιονομική διαδικασία, για παράδειγμα, τα έγγραφα ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούν να τροποποιήσουν τα κείμενα που φτάνουν σε αυτούς, μπορούμε απλώς να πούμε ναι ή όχι. Αυτό το άρθρο λοιπόν που προβλέπει το μόνο ναι ή όχι, θέλουμε να εξετάσουμε με την έκθεση του συναδέλφου Στρασκόφσκι από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Πώς ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Με μια σύγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Επιτροπή Ίντα και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων η οποία χρησιμοποίησε μια αναθεώρηση στον κανονισμό για να καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Η Επιτροπή Ίντα όμως δυσταρρυθμίστηκε όλος ιδιαίτερος από το έργο της Συνταγματικής Επιτροπής. Εκ παραλληλού, στη διάσκεψη πρόεδρων των Επιτροπών είχα εκφράσει και εγώ την ανησυχία μου για το σχέδιο έτσι όπως το είδα από τις εργασίες της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων. Γιατί η έκθεση Στρασκόφσκι εξακολουθούσε να μην αναγνωρίζει στις ειδικέ επιτροπές τη δυνατότητα να παρέμβουν μέσα σε μια τέτοια διαδικασία. Και αυτό το είδαμε και στη συμφωνία που τη λέμε DT, η διατλαντική δηλαδή, όπου οι κοινωνικέ προδιαγραφέ πώ λαμβάνονται υπόψη στι διαπραγματεύσει μια τέτοια συμφωνία είναι ένα θέμα που εμά βέβαια μα απασχολεί πολύ. Όμω δεν είχαμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε. Αυτό λοιπόν το είπα στην Επιτροπή Προέδρων Επιτροπών και όταν η ΙΝΤΑ δυσαρεστήθηκε και με τα αποτελέσματα τη Συνταγματική Επιτροπή, γι' αυτό αποφασίσαμε και εμεί να γνωμοδοτήσουμε επί της τροποποίησης αυτή που προτείνει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Επί της ουσίας. Ο συνάδελφος Τζαπαουρή από το ΕΛΚ ε, βοήθησε και καταλήξαμε νομίζω σε μια αρκετά καλή συμφωνία και ελπίζω ότι η ψηφοφορία θα αντικατοπτρίσει ακριβώς αυτή τη δυναμική. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για τρία προβλήματα. Τι λέει βασικά η ΑΦΚΟ. Λέει υπάρχει ένα πρώτο εγγραφό για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ναι ή όχι και μετά υπάρχει ένα ψήφισμα για να διευκρινιστεί αυτό το ναι ή όχι. Ο εισηγητής στην ΑΦΚΟ πρότεινε η σύσταση με την οποία λέμε ναι ή όχι δεν περιλαμβάνει αιτολογικές σκέψεις, μόνο την ίδια την ε, σύσταση και τα θεωρώντας. προτείνεται μια πολύ σύντομη αιτιολόγηση. Εγώ πρότεινα στον Σεφερή που συμφώνησε στο νομικό καθεστώς που θα είναι η αιτιολογική σκέψη που θα συνδέεται με την σύσταση να χρησιμοποιήσουμε το κοινό δίκαιο. Δηλαδή, εάν η αιτιολογική σκέψη δεν αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο τελικά θα έχει ψηφίσει η Επιτροπή, τότε ο πρόεδρος της Επιτροπής να μπορεί να ζητήσει αυτή η αιτιολόγηση, η οποία δεν θα συνάδει πια με τη σύσταση, να αποσύρεται. Το δεύτερο σημαντικό, και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, γιατί νομίζω ότι δεν ήταν ξεκάθαρο για μας στην αρχή, αυτό που προτείνει η Επιτροπή ΑΦΚΟ, εάν την ακολουθήσουμε, ακολουθήσουμε τον εισηγητή δηλαδή, θα σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορεί πια να απορρίπτει κείμενο το οποίο του υποβάλλεται για σύμφωνη γνώμη. Μόνο ναι θα μπορούμε να πούμε ή να αφήνουμε τα πράγματα ως έχουν. Και εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια άρνηση δημοκρατίας. Τι δημοκρατία είναι αυτή, γιατί εάν το κοινοβούλιο δεν θέλει να πει ναι, ε, πρέπει να έχει δικαίωμα να πει όχι. Αυτό όμως το οποίο σήμερα μας προτείνει η Επιτροπή Σταματικών Υποθέσεων είναι ότι μας απαγορεύει να πούμε όχι. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι αυτό το οποίο μας προτείνουν είναι ή που θα πείτε ναι ή που τα πράγματα παραμένω έχουν μέχρι να πιστείτε και να πείτε ναι. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό και εγώ προτείνω να διαγράψουμε όλη αυτή την αμφισημία, η οποία δεν βοηθάει και που προτείνει η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Και από ό,τι έχω καταλάβει, ο συνάδελφος Σαμπαόρη συμφωνεί και χαίρομαι γι' αυτό. Τρίτο. Κάτω από ποιες συνθήκες η δικιά μας Επιτροπή μπορεί να παρέμβει για να γνωμοδοτήσει σε μια τέτοια περίπτωση. Εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο τμήμα ή μάλλον στη μέση της συμβαστικής τροπολογίας που σας προτείνεται και όπου έχουμε συμφωνία με τον κύριο Ρή. Πράγμα το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Υπάρχει και η τροπολογία 7 που προτείνει ο κύριος Τσαμπορή, που νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή τροπολογία και η οποία λέει ξεκάθαρα ότι το επεξηγηματικό ψήφισμα και τη ολόγηση που θα ψηφιστεί πέρα από την σύσταση πρέπει να χρησιμεύει για να διευκρινίσει την εντολή και τις διαπραγματεύσεις. Ο εισηγητής είχε προτείνει στην αρχική του διατύπωση το ψήφισμα αυτό να μιλάει για τις διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή. Εγώ προτείνω κάτι προφορικά που λέει ότι το ψήφισμα αυτό πρέπει να αποτελεί τη βάση για την εντολή της Επιτροπής. Δεν λέμε ότι είναι η εντολή, λέμε ότι είναι η βάση της εντολής. Όπως το είχαμε δει και με την ψηφοφορία για την Διατλαντική Συμφωνία. Συγγνώμη που σας είπα ίσως περισσότερα από όσα περιμένατε σήμερα το πρωί τέτοια ώρα για θεσμικά ζητήματα, αλλά πάση περιπτώσει πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτά για να μπορούμε να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε επί της ουσίας. Είναι ξεκάθαρο αυτό ή θέλετε κάποια εξή. Παρακαλώ, Αλεχάνδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις σας και για την ενέργειά σας. Μπράβο, χαίρομαι βλέπω ότι οι ικανότητες του Κοινοβουλίου και τη επιτροπή αυτή βρίσκονται σε καλά χέρια. Ένα σχόλιο για την τροπολογία 7 των σοσιαλιστών. Ακριβώς αυτό το οποίο θέλαμε είναι να μπορούμε όπως και με τις κανονικές διαδικασίες να μπορούμε να δίνουμε την μάχη μας στην διάσκεψη των Προέδρων ώστε ως επιτροπή γνωμοδοτούσα να μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς. Οπότε βλέπουμε ότι το άρθρο 7, η οριζόντια ρήτρα, κυρία Πρόεδρε, για τα κοινωνικά ζητήματα, συστηματικά είναι κάτι που ξεχνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, σε τέτοιες περιπτώσεις, και είναι πολλές, πραγματικά πολλές κατά τη διάρκεια της εντολής μας, όπου τίθενται ζητήματα κοινωνικά, αν μη τι άλλο, να μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε με ξεκάθαρο τρόπο και με απόλυτη συνέπεια με τους κανόνες που ισχύουν. Πρόεδρος, ναι, ακριβώς. Άλλος κανείς, όχι, ωραία. Οπότε αργότερα θα έρθουμε στην ψηφοφορία αυτού του κειμένου. Στις τροπολογίες δηλαδή της Δεματικής Επιτροπής. Σημείο 14 τώρα. Η κυρία Ζέσκα όμως θα αντικαταστήσει τον εισηγητή μας τον κύριο Μάρτιν Κάσλερ. Πρόκειται για την εξέταση γνωμοδότησης. Το θέμα είναι γυναίκες μετανάστριες χωρίς έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Όσον αφορά λοιπόν τις γυναίκες μετανέστριες χωρίς έγγραφα, πρέπει να σας πω ότι η πλειοψηφία των γυναικών αυτών μετά από ένα χρονικό διάστημα έρχονται αντιμέτωπες με δυσκολίες και δεν έχουν τελικά τα κατάλληλα έγγραφα για να μπορούν να ζήσουν ή να δουλέψουν στη χώρα στην οποία βρίσκονται. Το θέμα αυτό λοιπόν των ε, μεταναστριών αυτών ε, των ε, παράτυπων και αντικανονικών οδηγεί σε φοβερές δυσκολίες και βρίσκεται εκτός ελέγχου. Οι γυναίκες αυτές και τα παιδιά τους είναι τα πιο ευάλωτα θύματα. Ιδιαίτερα όσοι έχουν επιζήσει εδώ οικογενειακής βίας, για παράδειγμα η προβλημάτων στην εργασία που δεν έχουν καμία προστασία. Τα θύματα μεταφέρονται, τους διώχνουν δηλαδή από τις χώρες τους εφόσον καταγγείλουν κάποια κατάχρηση. Γι' αυτό λοιπόν η γνωμοδότηση του κυρίου Κάστερ λέει ότι όταν υπάρχουν γυναίκες χωρίς έγγραφα ιδίω που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη, οι μητέρε, οι ανήλικοι ζητούν πρόσβαση στη δικαιοσύνη κλπ, τότε δεν θα πρέπει να δίνουμε σημασία μόνο στην παρατυπία τους, αλλά και στο καθεστώς του θύματος. Πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα υπέρ της προστασίας από τη βία, από την εκμετάλλευση και την διάκριση. η ανθρωπότητα και το στοιχείο του ανθρώπου πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο. Η γνωμοδότης λοιπόν του κύριου Κάστερ προορίζεται για την Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Οι μετανάστρες αντιμετωπίζουν πολλά νομικά και διαρθρωτικά εμπόδια, τα οποία τις δυσκολεύουν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η στέγαση, η νομική αρρωγή, η προστασία στους χώρους εργασίας η γνωμοδότηση ζητάει από τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν μέτρα για την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην αγορά εργασίας και να τις βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορούν να ασκούν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Η γνωμοδότηση ζητεί να θεσπιστούν ειδικέ μορφέ προστασία των ε, δεδομένων για τι γυναίκε που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα, οι οποίε ε, είναι θύματα, ώστε να μπορούν να καταφύγουν σε καταφύγε ιδρύματα υποδοχή γυναικών ή υπηρεσίε παροχή ε, συμβουλών δίνει γνωμοδότηση ιδιαίτερη σημασία στι γυναίκε χωρί έγγραφα, οι οποίε βρίσκονται σε κατάσταση δικαιοσύνη ή έχουν μικρά παιδιά. Χρειάζονται ειδική προστασία επίση για τα γέννητα παιδιά και πρέπει να έχουν νομικό δικαίωμα σε ιατρική μέρημνα, καθώ και δικαίωμα σε επιστοποιητικό γέννηση για το παιδί του, σύμφωνα με το άρθρο 7 τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είμαι σίγουρη ότι στην Επιτροπή αυτή υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων ότι πρέπει να φροντίζουμε για τις γυναίκες χωρίς έγγραφα. Αν μη τι άλλο, Μάρτιν Κάσλερ μου ζήτησε να σας πω ότι προσπάθησε να λάβει υπόψη του τις 1500 επιστολές που πήρε και είναι ανοιχτός σε οποιοδήποτε συζητήσεις και διάλογο που θα προκύψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Γιακονσάρη τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ συχνά μιλάμε για παράνομη μετανάστευση ή για παράνομους μετανάστες. Μα ένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να είναι παράνομος. Οπότε για να είμαστε σωστοί στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε δεν πρέπει να μιλάμε για παράνομους μετανάστες αλλά για μετανάστες χωρίς έγγραφα. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα και που οδηγεί σε πολύ σοβαρές κοινωνικές καταστάσεις έχει σαν αποτέλεσμα οι μετανάστες χωρίς έγγραφα να είναι εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο και στις κάτω και στη Φιλανδία. Εκεί γυναίκες που πάνε να γεννήσουν στο νοσοκομείο και που δεν έχουν έγγραφα, οι γυναίκες αυτές πρέπει να πληρώσουν 500 ευρώ εγγύηση πριν μπουν στο νοσοκομείο. Ε, όχι, δεν μπορεί να είναι αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δράσουμε και γι' αυτό είναι καλό που ζητάει η γνωμοδότηση αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι να δράσουν στους χώρους εργασίες, να ληφθούν διάφορα μέτρα για να προστατεύονται οι γυναίκες αυτές χωρίς έγγραφα. Το βασικό για μένα είναι στα πλαίσια αυτά να επενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μεταναστευτική μας πολιτική είναι κατακαιρματισμένη. Βασικά δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί. Και είναι η Ευρωπαϊκή Ακριβώς Επιτροπή εκείνη η οποία πρέπει να αλλάξει τα πράγματα. Οι γυναίκε, λοιπόν χωρίς έγγραφα δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και να το επαναλάβουμε. και στην Ολομέλεια πρέπει να το πούμε και πρέπει να συμπεριληφθεί στην πολιτική συζήτηση που γίνεται γιατί η οικονομική κρίση πλήττει όλους ιδιαίτερως τους πιο ευάλωτους και κυρίως τις μετανάστριες χωρίς έγγραφα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλο κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Η Τζιν Λάμπερτ. Σας ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για τη γνωμοδότηση αυτή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να τα πει κανείς όλα μέσα σε τόσο μικρό κείμενο όσο μπορούμε να προσφέρουμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχει και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας που αναφέρεται στους ανθρώπους που χρησιμοποιούνται ως οικιακή βοηθή αυτοί παγιδεύονται πολύ συχνά μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Ίσως πρέπει να επενθυμίσουμε και τα πράγματα που έχουμε πει για την πρόσβαση στην υγεία, για παράδειγμα, το είπε και η κυρία Γιακονσάλη, κυρίως για τις γυναίκες που περιμένουν παιδί, που είναι σε ενδιαφέρουσα ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στην φροντίδα για τις εγγύους και τα νεογέννητα. Γνωρίζουμε ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή αυτή. Λοιπόν, συμφωνώ με την γνωμοδότηση και θα υποβάλουμε τροπολογίες προς την ίδια πάντα κατεύθυνση για να εμπλουτίσουμε το κείμενο. σε ευχαριστούμε. Αναφερθήκατε στη σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Η σύμβαση αυτή άρχισε να ισχύει στις 5 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς, μόνο δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν επικυρώσει τη σύμβαση αυτή, η Γερμανία και η Ιταλία. Συνεπώς, τα μέλη της Επιτροπής μας, παρά τις δυσκολίες των κυβερνήσεων, ίσως θα έπρεπε να τους ε, ζητήσετε, να κινητοποιηθείτε δηλαδή και να ζητήσετε από τις κυβερνήσεις σας να την επικυρώσουν. Γιατί δεν το κάνουν, ρωτήστε τους. Γιατί δεν έχουν επικυρώσει ακόμα αυτή τη σύμβαση που για μας είναι τόσο πολύ σημαντική, γιατί τόσες χώρες δεν έχουν επικυρώσει. Άλλος κανείς θέλει το λόγο για αυτό το θέμα, όχι. Εκπρόσωπος της Επιτροπής. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Σύντομα, γιατί πρέπει και να ψηφίσουμε. Η κυρία Αρντοβίνα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, ναι. Θέλω να σας προσθέσω κάποια στοιχεία για τα διάφορα σημεία που αναφέρονται στη γνωμοδότησή σας. Πρώτα απ' όλα για την οδηγία 2009-52 που αναφέρεται σε ελάχιστες προδιαγραφές για κυρώσεις και μέτρα για τις περιπτώσεις ε, ατόμων που παράνομα βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να σας πω ότι πράγματι προσπαθούμε να αλλάξουμε την ε, οδηγία για του χρόνου. Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2011-36 για την πρόληψη και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπων και προστασία των θυμάτων στις χώρες μέλη, όπως ξέρετε, η προθεσμία έληξε τον Απρίλιο. Τώρα είμαστε λοιπόν στη διαδικασία αξιολόγησης της ενσωμάτωσης στην Εθνική Νομοθεσία. Κάνουμε και έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής εν του 2016. Όσον αφορά τώρα το σημείο 5 για την εκτεταμένη έρευνα που χρειάζεται για το πόσα άτομα βρίσκονται σε Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγγραφα παραμένει. Ίσως θα ήταν καλό να γνωρίζετε ότι όπως έχουμε ανακοινώσει κι αλλού, η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια μελέτη για τη διαφορά στο φύλλο, δηλαδή πιο συγκεκριμένα πόσες γυναίκες βρίσκονται στην κατηγορία αυτή χωρίς έγγραφα. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα να τα έχουμε σε ένα-ενάμιση χρόνο. Πρόεδρος, ε, η συγκήτρια. Θα τα μεταφέρετε όλα αυτά, έτσι, στο συντάκτη της γνωμοδότησης. Σωστά. Σωστά. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιώργη Συμφωνείτε κι εσείς, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ. Οπότε, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα εξεταστούν οι τροπολογίες στις 5 Νοεμβρίου εδώ στην Επιτροπή μας 25 Νοεμβρίου συμβαστικές τροπολογίες και την επόμενη 26 Νοεμβρίου δηλαδή θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Η Επιτροπή Γυναικών θα ψηφίσει στις 16 Δεκεμβρίου. Οπότε ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Όμεν Ράουτεν πρόκειται να μας ενημερώσει για τον τριμερή διάλογο, όμως δεν έχει έρθει ακόμα αυτό που έγινε χθε το βράδυ. Οπότε βάλετε αυτό το σημείο. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία και αρχίζουμε την ψηφοφορία. Σημείο 17 λοιπόν ψηφίζουμε πρώτα για την ε, νομοθετική έκθεση της συναδέρφου Σάρι Εσαγιά που είναι σχέδιο έκθεσης για τροποποίηση των οδηγιών 9258, 9285, 9433, 9824 και 2004-37 ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό 1272 κάθετος 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων. Πρόκειται για ένα νομοθετικό κείμενο λοιπόν που λιγάκι καθαρίζει το πεδίο. Κινητοποιήθηκε η συγγητριά μας με μεγάλο επαγγελματισμό. Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί τις τροπολογίες 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, όχι, καλώς. Οπότε, αρχίζουμε. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε 4. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε 5. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε 6. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε 7. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε 8 κατά υιοθετείτε. 9 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε, 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 15 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 16 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται, 17 υπέρ κατά αποχές 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Υιοθετούνται όλα λοιπόν, πρώτο εκτιμώντας, συμβασμός α, που παρουσιάζεται από δύο μάτς, υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Εκτιμώντας 5, συμβασμός β, από τις δύο ομάδες υπέρ κατά αποχές Υιοθετείται. 7. Τροπολογία 23. Άρκιν. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Ε, 24. Καταπίπτει. Και ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο του σχεδίου έκθεσης. Θα προσθέσουμε και μία ψήφο, ε. Δύο, γιατί δεν έχουμε κάρτα. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται το σχέδιο έκθεσης. 34, συγγνώμη, 34 ψήφι υπέρ. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Πάμε στο σχέδιο ψηφίσματος, νομοθετικού ψηφίσματος και ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Και τώρα θα πρέπει να επαληθεύσουμε αν θέλουμε να δώσουμε μια εντολή διαπραγμάτευσης στην εισηγήτρια και στην διαπραγματευτική ομάδα. Η διαπραγματευτική ομάδα αποτελείται από την εισηγήτρια της Άρια Σαγιά, εκπροσωπεί το ΕΡΚ, Όλε Κρίστιανσεν για τους σοσιαλιστές, Μαριάννα Χάρκιν από τους φιλελεύθερους, Καρίν Μαντέλη από τους πράσινους και ο Μακιντάιρ, η Ανθέα Μακιντάιρ από το ECR. Αυτή είναι η ομάδα διαπραγμάτευσης. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εντολή διαπραγμάτευσης με βάση το νομοθετικό ψήφισμα όπως το τροποποίησαμε, θα πρέπει τουλάχιστον 25 μέλη, 25 βουλευτές, να ψηφίσουν υπέρ. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την εντολή τώρα με ηλεκτρονικό τρόπο. Ξεκινάτε. Τη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Μπράβο κυρία ηγητρία. ψηφίσουμε το 18 ή έπρεπε τουλάχιστον. Αντίθετα σε όλους τους κανόνες όμως η κυρία Παπαδοπούλου μου ζήτησε να ψηφίσουμε τώρα τη δική της έκθεση. Έχει κανένα αντίρρηση? Όχι. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος Παπαδοπούλου. Πάμε λοιπόν στο σημείο 24. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη. Και για να κυλήσουν ομαλά οι εργασίες μας, κανονικά πρέπει να το πείτε τότε. Πάμε λοιπόν στο σχέδιο έκθεσης κυρίας Παπαδοπούλου. Είναι μια έκθεση γνωμοδότηση για την, προς την Επιτροπή ΛΥΠΕ. Είναι μια πρόταση οδηγίας για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, της σπουδέ στην ανταλλαγή μαθητών, την έμιστη ή πρακτική άσκηση, την εθελοντική εργασία και την ε, απασχόληση ως εσωτερική άμυστη βοηθή, ο ΠΕΡ. Άρθρο 1, σημείο α. ετροπολογία τροπολογία 21 της ηγήτρες υπέρ, κατά, πορχές απορρίπτεται. 22 της εισηγήτρες υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 94 καταπίπτει. Πάμε λοιπόν στο άρθρο 3, ε, σημείο F, κομπρομή G. Περ, κατά, αποχές υιοθετείται. Άρθρο 3, τροπολογία 96, Jean Λάμπερτ Μάλικα Μπενάρα Μπατού, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 3, σημείο E, συμβασμός H, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται. Ο ε, 99 καταπίπτει. Πάμε άρθρο 3, σημείο M, συμβασμό I, υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 31 της ηγετρίας υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 32 της ηγετρίας υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 33 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 σαρίσα για υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την 101 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 20 κατά, κατά ε, απορρίπτεται. Άρθρο 4 παράγραφος 2. Τροπολογίες 102, 103, 36 που είναι ίδιες. Τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείτε. Τροπολογία 104. Υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείτε. 37 της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ...38 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός J των δύο ομάδων υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Τροπολογία 40 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός K υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός L τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45, τροπολογία 45, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 109 δεν είναι παραδεκτή. Συμβασμός αίμα, δύο ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 47 της εισηγήτρες, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη 47. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. 16 πέρι 22 κατά. Δεν υιοθετείται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβιβασμός N δύο ομάδων υπέρ κατά αποχές υιοθετείται δύο τροπολογίες κατάργησης, 112 και 113, που είναι ίδιες, τις ψηφίζουμε μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός O, τριών ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 53, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 δεν είναι παραδεκτή. 115, 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 116. Ψηφίζουμε υπέρ, σε 116, κατά, αποχές, υιοθετείται. Άρθρο 12, παράγραφος 2, η 117, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα, θα ψηφίσουμε το συμβασμό π δύο ομάδων. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Δύο τροπολογίες κατάργησης, οι 119 και 120. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετούνται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 119 και 120. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 21 ψήφι κατά. Όχι, 19, 19 έκανα λαθο Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Άξιζε την επαλήθευση. 121 υπέρ. Κατά. Αποχέσιοθετείται. 124 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Συμβασμός Q υπέρ κατά άποχες υιοθετείται. Τροπολογία 57 της εισηγήτρες υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι περνάει αλλά θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας 19 υπέρ 20 κατά απορρίπτεται. Συμβασμός R Σοσιαλιστών και Λαϊκού Κόμματος υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται. 59 της εισηγήτρες υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά αποχές. Θα την επαληθεύσουμε την 60 ηλεκτρονικά. Ψηφίζετε. Όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 24 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. 128. Σαρίσα για υπέρ, κατά, άποχες. Υιοθετείτε. 61 της ηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 62-63 είναι μη παραδεκτές. 129 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε την 129 ψηφίστε ηλεκτρονικά τώρα πέρας ψηφοφορίας «20 υπέρ, 19 κατά, υιοθετείτε». 130, σάρι σαγιά, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 131 της φυγής ηγήτριας υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 64 της ηγήτριας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 Ισαΐα υπέρ. 132 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση της 132. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας φοφορίας 19 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Πάλι είχατε δίκιο. Άξιζε η επαλήθευση. 133. Χίρς υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 134. Την 133 θέλετε να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζετε τώρα. Πέρας προφορίας. 20 υπέρ, 19 κατά, υιοθετείτε. 134, σάρισα για υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 135, υπέρ, κατά, αποχές, επαληθεύουμε. Ψηφίζετε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 19 κατά, υιοθετείτε με την ίδια πλειοψηφία. 136 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 137 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Υπάρχει κάτι στον κατάλογο ψηφοφορία που δεν καταλαβαίνω. Να ψηφίσουμε λέει πρώτα τον συμβασμό S υπέρ. Κατά απόχε. απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίσουμε την 65 της Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Ψηφίσαμε λοιπόν τον συμβασμό S, έτσι. Ξαναψηφίζουμε και επαληθεύουμε την τροπολογή των συμβιβασμό S. Έτσι. Ψηφίστε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 31 ψήφι ΠΕΡ, 8 κατά, υιοθετείτε. Πάμε στο συμβιβασμό τι τελικά. Υπέρ. Κατά αποχές Υιοθετείτε. Σεβασμός γιου, υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. Εκατόν Σάρια Σαγιά, υπέρ. Α, ο διορθώνει 146, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 147 καταπίπτει. Συμφωνεί η Συμφωνεί η 69. Η 69 της συγκήτριας είναι απαράδεκτη. Ψηφίζουμε τώρα μαζί την 148, 149, 150 και 151 της Jean Lambert. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Δεν τροποποιείται το άρθρο 25. 152. Υπέρ. Κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. φανταζόμουν θα το ζητούσατε εσείς το, το, το να επαληθεύσουμε την 152. Τώρα ψηφίστε λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 19 κατά. Υιοθετείτε. Κλασική πλειοψηφία σήμερα το πρωί, μια ψήφος διαφορά. Πάμε την, στην 72. Υπέρ. Της 72. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. Ψηφίζουμε την 155 τώρα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι υιοθετείτε, αλλά επαληθεύουμε. Ψηφίζουμε την 155. 20 υπέρ 19 α, κατά κλασικά. Για 73 αποσύρεται, για 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Δεν 77 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 155. Σαρίσα Αγιά. Κατά. Α, όχι, λάθος έκανα 158, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τις αιτιολογικές σκέψεις. 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 3, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός α. Σοσιαλιστών και ΕΛΚΑ υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 6 Τις ηγήτρες υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Την 79 δεν την ψηφίσουμε. Την 80 έδωσε σε θέλω. Την ψηφίζουμε. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός B. Δύο ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 8 της εισηγήτριας. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 12 11. Επαληθεύουμε την 11 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ναι. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 21 κατά. Δίκιο είχατε. Απορρίπτεται 12 υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείτε. Συμβασμό C, τριών ομάδων υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείτε. 28 Συγγνώμη, εκτιμώντας 28, ε, τροπολογία 84 απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 14 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 15 της ηγήτριας κατά αποχές απορρίπτεται. 87. «87» της Νάντια Χίρς, υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. Συμβασμός D των δύο ομάδων, υπέρ, κατά, απόχες, υιοθετείται. 16. Υπέρ, κατά, απόχες, επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Καλύπτεται η 17, άρα ψηφίζουμε τη 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός Ή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και πάμε τώρα. Θέλετε να επαληθέσουμε το 92. Να την Ψηφίστε ηλεκτρονικά την 92. Ψηφίσαν όλοι πέρασε τη φοφορίες. 17 υπέρ 21 κατά απορρίπτεται. Χωρίς καμία αποχή. Συμβασμός F των δύο ομάδων υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Ψηφίζουμε το σύνολο ηλεκτρονικά τη γνωμοδότησης. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. 30 υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή. Μπράβο στην εισηγήτρια. Είμαστε πάντα με τη σειρά στις ψηφοφορίες και φτάνουμε στο σημείο 18 έκθεση Κόζα. Πρόκειται για σχέδιο που ετοιμάζουμε. Α, όχι, εμείς είμαστε αρμόδια Επιτροπή επί της ουσίας. Πρόκειται για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Έχουμε και γνωμοδότηση από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ελευθερία του Πολίτη. Παράγραφος 1. Τροπολογία 17. Σέντερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. 17. Σρέντερ. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. Μετά την παραγραφό 1, 18 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ένα β από τρεις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, 22 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, 24, Σρέντερ, με προφορική τροποποίηση της συγκήτριας, υπάρχει αντίρρηση, όχι, ψηφίζουμε λοιπόν τροποποιημένη τροπολογία, 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3, παράγραφος 2 της Επιτροπής Λίμπη κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος... Α, να αλλάξουμε για την παράγραφο για το 2 της Λίμπε υπέρ. Πέρα στις φοφορίες 20 υπέρ, 16 κατά, 2 αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη της Λίμπη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, συμβαστική γάμα από 4 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Σρέντερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αλλά αν θέλετε να επαληθεύσουμε, να επαληθεύσουμε. Όχι, εγκρίνεται, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Καλά, να επαληθεύσουμε. 27. Σρέντερ, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική δέλτα τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29. Άνταμ Κόζα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Καλά, θα επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Λίμπε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Με ώρα κλειβέτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Τροπολογία 30. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της φοφορίες. 18 υπέρ, 20 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 31, κλειβέτη. Υπάρχει προφορική τροποποίηση. πρέπει να σηκωθούν τρία χέρια για να αντιταθούν στην προφορική τροποποίηση. Τότε δεν εγκρίνεται. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 31, κλειβέτη, ως έχει, χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά αποχές η 31 εγκρίνεται. Τροπολογία 32, κλειβέτη, με προφορική τροποποίηση. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν με την τροποποίηση την τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολίγια 33. Κλειβέτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Λασλό Σουζάν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Κλειβέτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38, κλειβέτη, με προφορική τροποποίηση του συντάκτη. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Κύριε Κοζά, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ίσως ε, πήγατε πολύ γρήγορα, αλλά για την τροπολογία 35 θα ήθελα να την αποσύρω. Δεν μπορούμε λοιπόν να την ψηφίσουμε την τροπολογία 35, επειδή ο συντάκτης την απέσυρε. Κύριε Σιγητά, σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε, αλλά εγώ δεν είπα 35, αφού είχε αποσυρθεί ακριβώς, για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα δεν το ανέφερα καν, να το πω, 35 και 37 έχουν αποσυρθεί, γι' αυτό και δεν τις έβαλα σε ψηφοφορία. Τώρα αυτό που λέμε είναι, έχει κανείς αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση της τροπολογίας 38. Είναι από τον ίδιο το συντάκτη, ε, τώρα Κλειβέτη. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροποποίηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 38 τροποποιημένη. Α, κύριε Κοζά πάλι, παρακαλώ. Είμαι κατά, κατά, εκ μέρους της ομάδας μου, κατά. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Είμαι κατά της προφορικής τροποποίησης, το λέω εκ μέρους της ομάδας μου. Ωραία, άρα ψηφίζουμε την τροπολογία 38 στην αρχική της μορφή, υπέρ της 38, χωρί την προφορική τροποποίηση. Κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε παρακαλώ. Τροπολογία 38, μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορίας. 15 υπέρ, 19 κατά, 4 αποχές. Απορρίπτεται. 39. Κλειβέτη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40. Ντανιέλ Φαντερστούπ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41. Φαντερστούπ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Λάσλο Ζουρζάν. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολίγη 43, κοζά, υπέρ. Να επαληθεύσουμε για την 42. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά 42. Ψηφίσατε όλοι, πέρες προφορίας. 22 υπέρ, 16 κατά, Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Εγκρίνεται. 43 τώρα. Κοζά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 Αντάμ Κοζά. Με προφορική τροποποίηση του ίδιου του εισηγητή. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε συνεπώς την τροπολογία 44 τροποποιημένη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίες. 21 ψήφοι υπέρ, 17 κατά. Η συμβαστική ε εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F σιγματά δύο ομάδων υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι υπέρ της συμβαστική F σιγματάφ Εγκρίνεται. Στη συνέχεια, τροπολογία 47. Λασλό Σιουζάν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G, Z, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 3, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50, κλειβέτη, με προφορική τροποποίηση. Να έχετε αντίρρηση, όχι, ψηφίζουμε με τροπολογία υπέρ. Μα έχουμε ήδη αρχίσει την ψηφοφορία. Παρακαλώ, κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Είμαι κατά της προφορικής τροποποίησης στην 50. Καλώς, άρα ψηφίζουμε για την 40 πάλι. Τροπολογία 50 λοιπόν, χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ. κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 50. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51. κίνκα Κόντς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λίμπε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ λέει η πρόεδρος. Α, όχι, λείπει μια σελίδα, κάτι δεν πάει καλά. Όχι, όχι, όχι, μπέρδεψα τις σελίδες μου, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Μετά την παράγραφο 6, 16. Είμαστε στην Λίμπε 9, υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 52, κόζα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Κλειβέτη με προφορική τροποποίηση που προτείνει ο εισηγητής. Αντιρρήσεις για την προφορική τροποποίηση. Όχι, από ό,τι βλέπω. Οπότε ψηφίζουμε τροπολογία 53 με την τροποποίηση υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια τροπολογίες 54 και 55 καταπίπτουν και φτάνουμε στις αιτιολογικές αναφορές. Εδώ είναι πιο περίπλοκο όμως τα πράγματα. Αιτιολογική αναφορά. Υπάρχει μία που μοιάζει πολύ με τη σκέψη. Εν πάση περιπτώσει, το προτείνει ως αιτιολογική αναφορά και ζητάει κατά τμήματα ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα του κειμένου που για μένα θυμίζει το λογική σκέψη, ε, γιατί λέει λαμβάνοντα υπόψη το άρθρο 1 της ε, Χάρτας ε, Θεμελιδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ειδική μνήμα στο απαραβίαστο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χωρίς τη συνέχεια που λέει που αποτελεί ένα οικομενικό ανθρώπινο δικαίωμα. Εγώ είμαι υπέρ της προφορικής τροποποίησης, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε με την αιτιολογική αυτή αναφορά είναι ότι δεν μπορεί να κάνει μία αξιολόγηση. Πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς μόνο, να αναφέρεται σε κάποιο κείμενο, σε κάποιο νόμο. Γι' αυτό και βγάζουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι της πρότασης του συγητή, που αποτελούσε μια εκτίμηση, έκανε μια αξιολόγηση του δικαιώματος αυτού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυσκολία εδώ. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Το πρώτο τμήμα του ένα το Αντάμ Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, δεύτερο τμήμα. Και εδώ υπάρχει προφορική τροποποίηση του ίδιου του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου αυτού πρώτα απ' όλα για την προφορική τροποποίηση. Υπάρχει κανείς που έχει αντίρρηση με την προφορική αυτή τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις, άρα δεν προφοράει Άρα το υπόλοιπο δεν είναι αποδεκτό. Συνεπώς τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 2 του Σύριο κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, η τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί. Και ερχόμαστε στην συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 κλειβέτη υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε επαληθεύουμε τροπολογία 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. 21 ψήφι υπέρ, 17 κατά. Η τροπολογία 5 εγκρίνεται συνεπώ. Τροπολογία 6 κοζά υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο σίγμα ταφ, F, τροπολογία 7, Ελίζα κατά καταπίπτει, το ίδιο και η 8 και η 9 και η 10. Οπότε ερχόμαστε στην ε, σκέψη Z, G, Ελίζα Μπερσέτερ, υπέρ, τροπολογία 11. Κατά, αποχές θα επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε τροπολογία 11. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. 18 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην αλλογή σκέψη H 13 δεν την ψηφίζουμε και δεν εγκρίθηκε 51 και πάμε στην τροπολογία 14, τσάπα όρη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ιώτα, μάλλον Άι, δηλαδή θήτα. Εδώ καταπίπτουν όλα. Ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία λοιπόν. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν ε, το τέλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επειδή πρέπει να σας πω η σημερινή ψηφοφορία έγινε όπως έγινε, πρόκειται για τροπολογίες ε, για τις οποίες είχαμε συμφωνήσει, προφορικές τροποποίησεις που ήξερα ότι θα υποστήριζε. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω ότι άλλαξαν τα δεδομένα. Εδώ με εκπλήσει η ψηφοφορία. Οι σοσιαλιστές τελικά αποφάσισαν να μην υποστηρίξουν την έκθεση αυτή. Και γιατί. Θα σας δώσουμε μια εξήγηση γιατί για μας πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση. Πολλές τροπολογίες υποβλήθηκαν. Δεν είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Προσπαθήσαμε βέβαια να δουλέψουμε με ανοιχτό πνεύμα αλλά δυστυχώς θα καταψηφίσουμε. Δεν θα υποστηρίξουμε την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, καλώς. Ε, άλλη επεξήγηση ψήφου υπάρχει πριν ψηφίσουμε. Ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο της τροποποιημένης έκθεσης του κυρίου Κόζα ηλεκτρονικά. Έτσι, ψηφίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της προφορίας. 17 ψήφοι υπέρ, 19 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται η έκθεση Κόζα. Συνεπώς δεν θα γνωμοδοτήσουμε, μάλλον διορθώνει πρόεδρος, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν εγκρίναμε την έκθεση πρωτοβουλίας του Άνταμ Κόζα για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την οδηγία του Συμβουλίου που αναφέρεται στην ίση μεταχείριση, στην απασχόληση και την εργασία. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο οποίος εννοείται ότι θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η εξέλιξη αυτή με εκπλήσει. Χτες, στη συζήτηση που έγινε εδώ, ακούσαμε ότι υπήρξε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Αλλά σύμφωνα με τους σοσιαλιστές, από ό,τι φαίνεται, δεν χρειάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει τη σημασία που δείχνει σε αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία κατά αποτελεί μια διάκριση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Αλεχάντρο Θέρκας. Αλεχάντρο Θέρκας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πρόθυμοι να ψηφίσουμε την έκθεση του κύριου Κώστα. διότι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που αναφέρθηκε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς η καταπολέμηση κάθε τύπου και μορφής αδιακριτικής μεταχείρισης. Το πρόβλημα είναι όλοι γνωρίζουμε όταν υπάρχει μια τέτοια έκθεση ότι πρέπει να φουγκράζεται, να ακούει και να σέβεται τις άλλες ομάδες και να έχει ένα διάλογο ανοιχτό με τις άλλες ομάδες και να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια με τις άλλες ομάδες και δεν μπορεί στη δική τους διακριτική ευχαίρεια να πει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τροπολογία χωρίς καμία δικαιολογία και καμιά βάση. Είναι ένας κανόνας που ε, έχει διαραγεί σε αυτή την έκθεση. Πάντα η ομάδα μας ήταν ανοιχτή σε τέτοιου είδους συμβιβασμούς. Όταν όμως κλείνει η πόρτα επανειλημμένα σε τέτοιες προσπάθειες υπάρχει ένα όριο. Κάποτε λέει κάποιος «Ε, φτάνει πια, δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί αυτό. Euh, Elisabeth Καταρχήν λοιπόν για το ότι ήταν μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλία που είχε την ιδέα πριν από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει κίνητρα και προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δική της έκθεση. Δηλαδή ήταν πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου που τώρα πέτυχε έτσι. Λοιπόν, η Επιτροπή παρόλα αυτά θα καταθέσει, θα υποβάλει τη δική της έκθεση και μπορούμε να αντιδράσουμε με δεύτερη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας εμείς. Διαδικαστικά αυτό, δεν, χάσα, δεν χάθηκε τίποτα. Με, μπορούμε και με μια ερώτηση στην Ολομέλεια να εξετάσουμε αυτά τα θέματα σε σχέση με την έκθεση της Επιτροπής. Για την ουσία της έκθεσης, το είπα χθε προσεκτικά και το ανέφερα, βρήκα και εγώ ότι δεν πήγαν πολύ καλά, δεν πήγαν εξαιρετικά οι διαπραγματεύσεις. Οι προτάσεις άλλων ομάδων δεν ελήφθησαν υπόψη. Και σε ένα πολύ ουσιώδη συμβιβασμό, τι έγινε, ο συμβιβασμός, δηλαδή το αίτημα της ομάδας αντιστράφηκε στο αντίθετο. Χθες είπα ήδη ότι θα δούμε σε σχέση με την ψηφοφορία αν μπορέσουμε στο τέλος να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση. Και επειδή πήγε ακόμα χειρότερα η ψήφιση ή η ψηφοφορια από ό,τι διαπραγματεύσεις δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν υπεψηφίσαμε την έκθεση. Και μπορώ να πω ότι είναι κρίμα, είναι βλάβη, κρίμα για το κοινοβούλιο αυτό. Βλάφτηκε το κοινοβούλιο, διότι ήταν πολύ μη ισόρροπη αυτή η έκθεση και δεν αναφέρε και δεν αξιολόγησε με τον ίδιο τρόπο όλους τους λόγους και τα αίτια της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Euh, άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Θέλει κανένας άλλος να εξηγήσει την ψήφο του. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς η Επιτροπή μας δεν μπορεί να πάρει θέση όπως το επιθυμούσε και όπως και οι συντονιστές ε, ήθελαν, είχαν εκφράσει την επιθυμία να εκφράσουμε, να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας αλλά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εξού και η σημασία του να δουλεύει κανείς μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας, ούτω ώστε να ξεκαθαρίζουμε ποια είναι τα ουσιώδη για μας και να μπορούμε να περνάμε τις θέσεις μας. Ο καθένας σας συνάγει τα συμπεράσματά του. Πάμε στο σημείο 19. Που αφορούν Σημείο 19 αφορά την ε, συνεισφορά μας στην τροποποίηση του άρθρου 81 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Παρα... Άρθρο 81, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1. Έχουμε ε, τον συμβασμό α εδώ Από δύο ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 5. Τσαμπά πέρι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ, παρακαλώ, ακόμα μια φορά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 5. Ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 15 κατά, μία αποχή. Έχετε δίκιο, υιοθετείτε. Τροπολογία 6, που είναι συμβατή με την 5 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά απόχες υιοθετείται η τροποποιημένη τροπολογία 7 με την προφορική τροπολογία. Τώρα έχουμε την τροπολογία 8 του Θέρκας. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Σας ευχαριστώ για την ψηφοφορία και πάμε στο σημείο 20. Θα ψηφίσουμε την έκθεση Πρωτοβουλία του Φιλίπ Μπουλόν. Τα μπέρδεψα. Όχι σχέδιο γνωμοδότησης. Για τη νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης, για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας. Στην παράγραφο 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός Α, α, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 6 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 7. Νταρντέν, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 8. Στάινρουκ, υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 9. Ίδιου εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός B. Τριών ομάδων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Τροπολογία 17. Σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας Darden χωρίς τη λέξη massively. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Ποιος είναι υπέρ της προσθέκη της λέξη massively, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 18. Υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείτε. 19. Υπέρ, κατά, άποχες, υιοθετείτε. Συμβασμός C, τριών ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 24 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 26 σύπερ υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα επαληθέσουμε ηλεκτρονικά την 26. tout le a le vote est clos. 18 υπέρ, 18 κατά. Απορρίπτεται. 27. Καρή Μαντελή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 28. Θέλετε να επαληθεύσουμε την 27. Να την επαληθεύσουμε. Υπέρ. Ή μάλλον λάθος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. 17 υπέρ, 17 κατά. Απορρίπτεται. Χρειάζονται λοιπόν σήμερα οι 28. Μπιργκίτ Σίπελ. 29. Ρέγνερ και 30. Δαρντέν είναι ταυτόσημες, τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, θα την επαληθεύσουμε και, αυτήν, και αυτές. Πέρας ψηφοφορίας. 18-18, η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται, απορρίπτονται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έχουμε αντίστροφη πλειοψηφία. Α, πρέπει να επαληθεύσουμε την 31. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, 19 υπέρ, 17 κατά. Υιοθετείτε. 32 υπέρ, κατά, αποχές. Υιοθετείτε. 33 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 34 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 35 υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. Συμβασμός D. Τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείτε. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Να ψηφίσουμε τις υπόλοιπες μαζί. Ωραία. Τη 40, 41, 42, 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετούνται. Ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 33 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή, Συγχαρητήρια. Πάμε στο 21. Σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή. Είναι και για την Επιτροπή Γιούρι για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση των νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών επί της άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Είναι θέματα επιτροπολογίας στην ιδιόγλωσσά μας. Τροπολογία 1, με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας της τροπολογίας. Είναι γλωσσική η αλλαγή. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1 πώς τοποθε... ε, τροπολο... τροποποιήθηκε, υιοθετείται. Συμβασμός A, δύο ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 6, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 7, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. On a pu voter, le vote est clos. 17 pour. 17 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Καταπίπτει. 8. Υπέρ κατά αποχές. 9 de Nadia Hirsch qui est pour, euh, qui est contre. Υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε. Την 9 τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ. 16 κατά. Υιοθετείτε. Ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότησης. Ψηφίζετε. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Θετείτε. Και πάμε τώρα στο 22, σημείο 22, για να ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης της Birgit Σίπελ για την Επιτροπή Ήτρε επί της έκθεσης του κ. Φρανκ Προύστ. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας για το σχέδιο δράσης για την βιομηχανία που τη θέλουμε ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη στην Ευρώπη. Μιλάμε για το ΚΑΡΣ 2020. Ψηφίζουμε το συμβασμό A. Τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές Υιοθετείτε. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Κορνέλισεν. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 1 όμως. Ποιο είναι υπέρ του δεύτερου τμήματο τη τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Τα έχετε λίγο, έχετε λίγο χαλαρώσει, έτσι. Πρέπει να το επαληθεύσουμε αυτό το σημείο. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 1 της, της κυρίας Κορνέλισεν. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 1. Ψηφίζεται. 17 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. Την 6, 7 και την 8 μαζί, θέλετε. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. Παράγραφος 2, συμβασμός B. Υπέρ, κατά αποχές υιοθετείτε. 12. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 13. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείτε. 14. θέλει τη διαγραφή. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός C. Τεσσάρων ομάδων. Υπέρ κατά αποχές. Υιοθετείτε. Δεκαεννιά. Υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Τη 19. Πέρας ψηφοφορίας, 20 υπέρ, 17 κατά. Υιοθετείται 19. 20 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Συμβασμός D τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός Ή τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 26 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Εφα, συμβασμός F4 ομάδων υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός G. Τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 34 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ 17 κατά Υιοθετείτε. 39 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 40 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 41 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 42 υπέρ κατά αποχές παληθεύουμε τη 42 Πέρας ψηφοφορίας. Δεκαεφτά υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της νομοδότης ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορία. 34 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια, κυρία Σίπελ. Και φτάνουμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Α, λάθος. Λέει πρόεδρος. Πρώτη τελευταία ψηφοφορία. Σημείο 23. Σχέδιο γνωμοδότησης της Φρανσουάς Καστέξ για την Οικονομική Επιτροπή. Η συνοραμών είναι ο Τρεμόσα και πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν την παράγραφο 1. Έχουμε τροπολογία 11 της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Από τέσσερις πολιτικές ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 τη εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε. Τροπολογία 12. Μπορείτε να ψηφίσετε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική σε γάμα από 4 ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 Μπουλό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 Καστέξ υπέρ, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. 23. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις 19 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά. Συμβαστική ε τριών ομάδων υπέρ κατά απέ. Τροπολογία 25. Μπούλον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Μπουλόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30, Μπενιόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31, υπέρ, καστέξ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε για τροπολογία 31. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοβορίας. 18 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική G, Z, από τέσσερις ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36, Κορνέλισεν, υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε. 36, ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Αλεχάνδρο Σέρκα υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική H. Ήτα τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Κοστέλο υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Α. Συμβαστική Α. Τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Κάζα. David Κάζα. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Καστέξη Σιγήτρη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. David Κάζα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. David Κάζα. Αποσύρθηκε. Ψηφίζουμε το σύνολο. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγητριά μας. Και ε, τις ευχόμαστε καλή επιτυχία για να επιβάλλει όλες αυτές τις απόψεις στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Κυρία Μπάουερ, εσείς τώρα. Όταν θα φτάσουμε στην ψηφοφορία του σημείου 25 του σχεδίου γνωμοδότησής σας, θα πάρετε τότε το λόγο. Είναι για την Επιτροπή Γυναικών και αφορά την έκθεση της κυρίας Γιάροκα που είναι έκθεση πρωτοβουλίας για τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης τον Ρωμά. Η συγγήτρια, παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως υποσχέθηκα και χθε όταν συζητήσαμε τους συμβιβασμούς, έγινε η προσπάθεια να βρούμε τις πιο κατάλληλες λύσεις όσον αφορά τις διατυπώσεις των συμβιβαστικών προτάσεων μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δυστυχώς πολύ, με πολύ καθυστέρηση ήρθαν απαντήσεις όσον αφορά το συμβιβασμό ΒΑ. Η τελευταία, ο τελευταίος έλεγχος μπόρεσε να γίνει δυστυχώς μόνο σήμερα το πρωί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να δεχθείτε την επεξήγησή μου, την τοποθέτησή μου, με τροποποίηση του BA, με κάποιες διατυπώσεις που θέλω να αναφέρω. Επίσης παρατηρεί ότι όλο και περισσότερο διακοπή χωρίς μικρόφωνο. Read something, just tell us where we are. Πείτε μας πού βρισκόμαστε, αντί να μας διαβάσετε κάτι. Ποιος... You know, you are in your text, we are not. <laughs> Ποιος συμβιβασμός, σε ποια σελίδα. Συμβιβασμός C. Προσθήκη. Μετά κοινωνικό αποκλεισμό λέμε και τοποθετούμε αυτά που πήραμε από την BA ως διατύπωση. Θέλω να σας το διαβάσω. Τέταρτη γραμμή παρατηρεί περαιτέρω ότι η αυξημένη γνώση για τον πολιτισμό των Ρωμά από πλευράς των καθηγητών ή δασκάλων βοηθά να περιοριστεί, να αναχαιτιστεί η περιθεωριοποίησή τους. Και νομίζω ότι μπορεί αυτό να είναι συνδεκτό και να ενταχθεί εδώ. Και στο συμβιβασμό ΑΕ κάπως διατυ... Ε, αλλάξαμε τη διατύπωση από αρνητική χρειά που είχε σε θετική απόχρωση στη τρίτη γραμμή. Κάνουμε λόγο για καλύτερη απασχολησιμότητα αντί ισχνή απασχολησιμότητα. Υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης αντί χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης και καταπολέμηση της περιθωριοποίησης, δηλαδή των διακριτικών, της διακριτικής μεταχείρισης. Ζητούμε δηλαδή να αναλυφθεί η δράση. Λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό, είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο, κάτι έκτακτο. Δεν είχαμε άλλη δυνατότητα όμως, διότι οι πρώτες τοποθετήσεις και ανταποκρίσεις σε σχέση με αυτές τις προτάσεις ήταν τα μεσάνυχτα μόλις. Ευχαριστώ. Πολλές καινοτομίε έχουμε κάνει σήμερα. Έχουμε αλλάξει την ημερήσια διάταξη εν μέσω της ψηφοφορίας, έχουμε απορρίψει μια έκθεση πρωτοβουλίας και τώρα αλλάζουμε και τις συμβαστικές τροπολογίες εν μέσω της ψηφοφορίας. Μα πού πάμε τέλος πάντων. Χρειάζεται κανείς διευκρίνηση για αυτά που για τις συμβαστικές τροπολογίες. Μαριάν Χάρκιν, για τις τροποποίησεις που προτείνει η συγκήτρια. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Μπάουερ. Στο συμβιβασμό, ε, είπατε ότι αντικαθιστούσαμε το που για την απασχολησιμότητα, ισχνή απασχολησιμότητα, με την λέξη καλύτερη απασχολησιμότητα. Αυτό δεν είπατε. Όχι και αντικαθιστούμε το χαμηλή με το υψηλή απασχολησιμότητα. Εντάξει, αυτό δεν είπατε. Αν επιτρέπετε κυρία Μπάουερ, όσον αφορά την ισχνή περιορισμένη απασχολησιμότητα που επαναλαμβανόταν στην τρίτη γραμμή, στην τρίτη γραμμή αλλάξαμε και είπαμε για καλύτερη δυνατότητα απασχόλησης, υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης. Από την πρώτη στην τρίτη γραμμή υπάρχει αυτή η αλλαγή διατύπωσης στην ορολογία. To, uh, be. Για το κείμενο όπως θα ήθελε η συγγήτρια να ψηφιστεί. Συζητάμε την τροπολογία ε, έτσι. Λοιπόν, υπογραμμίζει ότι η ισχνή απασχολησιμότητα χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή 2, 4, 5, 6, έκτη γραμμή. Στην έκτη γραμμή λοιπόν θα ήταν στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη ε, άρα ότι θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη καλύτερη απασχολησιμότητα, υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και καταπολέμηση των διακριτικό, της διακριτικής μεταχείρισης και στα σχολεία και στην αγορά εργασίας. Τα υπόλοιπα χωρίς αλλαγές. Αυτό είναι εντάξει, βαίνει καλός με όλους. Εγώ νομίζω βαίνει καλός και είναι αποδεκτό. Since we are uh, Αλλά μια και έχουμε καινοτομία νομοθετική με αυτή τη δράση σήμερα, ίσως έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Και είναι ικανοποιημένη η συγκήτρια με αυτό. Με τον ίδιο τρόπο να δούμε τώρα την τροπολογία C, να την συζητήσουμε. Και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε πάλι στο κείμενο. Σωστό αυτό, ναι. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Θα είχαμε από κειμένου στην έκτη στις έξι πρώτες γραμμές χωρίς κάποια τροποποίηση, μετά αποκλεισμό και μετά θα προσθέταμε ως προσθήκη παρατηρώντας περαιτέρω ότι η αυξημένη γνώση από πλευράς δασκάλων για τον πολιτισμό των συγκάνων βοηθά να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση και γι' αυτό καλεί τα κράτη-μέλη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπλα μπλα μπλα όπως θα έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, εντάξει, είναι όλα ξεκάθαρα. Ωραία, είναι ευχαριστημένη η συγκίτρια γιατί παρακάψαμε όλους τους κανόνες. Ψηφίζουμε. Αλλά προσοχή, ε, μην αποτελέσει νομολογία, γιατί τότε η γραμματεία δεν θα μπορεί πια να δουλεύει. Και θα ζητήσουν όλοι να φύγουν από την Επιτροπή μας και να πάνε σε άλλη. Λοιπόν, τροπολογία αριθμός 1. Ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική άλφα, τροποποιημένη, από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, κύριο ακόμη υπέρ, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, σάρισα για υπέρ, κατά, άποχες. Θα επαληθεύσουμε. Τροπολογία 9, εσαγιά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορίας. 16 υπέρ, 18 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10, κλειβέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Κλειβέτη. Με προφορική τροποποίηση. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροποποίηση. Όχι. Ψηφίζουμε την 11 τροποποιημένη υπέρ. Κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα προφορίας. 18 υπέρ, 18 κατά. Καμία αποχή. Απορρίπτονται οι 11. Ό,τι σχόλια έχουν οι πάλι εδώ πέρα, παρακαλώ εκτός εθούσης γιατί ενοχλείτε με την ψηφοφορία. Μην μιλάτε τόσο δυνατά. Κύριε Ρή, κάθε φορά προσθέτω δύο ψήφους. Ναι. Για τους σοσιαλιστές. Γιατί είναι οι σοσιαλιστές που δεν έχουν τις κάρτες τους, γι' αυτό τους προσθέτω δύο ψήφους. Τώρα, 12. κίνγα Κόντσιπερ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Με προφορική τροποποίηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ωραία, ψηφίζουμε τροπολογία 13 τροποποιημένη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 κοινά κόντς υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 κόντς υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β από 4 πολιτικές ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β Α από το ΕΛΚ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική εα από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21, King Cons. Διαγραφής υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 23, King Cons υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 ζωλίγου Μπεναμιάς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 Κιγκακόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 Κιγκακόντς υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Τροπολογία 26. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες. 7 και 2 ίσον 19 υπέρ, 16 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται 26. Συμβαστική γάμα σε 4 ομάδων. Παράγραφος 5. Συμβαστική Σ γάμα όπως παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική Δ Δέλτα της ονομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Κλειβέτη υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται 31. Τροπολογία 32 και υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Κλειβέτη. Α, όχι, να επαληθεύσουμε τη 32 λέτε πρώτα. Εντάξει. Ψηφίστε παρακαλώ. 32. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις φοφορίας. Δεκαεννέα υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. Το 33 κλειβέτη Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. 33. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της φοφορίας. 19 υπέρ, 17 κατά, η ίδια πλειοψηφία, εγκρίνεται. Παράγραφος 6 τώρα. Συμβαστική ε. Η τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 38 εισαγιά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 κίνκα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική εύσημα τάφ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική G, Z, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H, Ι, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54, σαρίες αγιά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55, μεναμιάς υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56, κινακόντς υπέρ, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. 56. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. 19 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 57, εισαγιά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 58, μια υπέρ, Α, λάθος, λάθος. Καταπίπτει αυτή. 59, King Acons. Υπέρ. Μαζί. Μπλοκ. 59, 60, 62, 63, 64, 65. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν όλες αυτές τις τροπολογίες μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη γνωμοδότηση ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της 3 32 υπέρ, 3 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τώρα, τελειώσαμε με την ψηφοφορία, αλλά στο σημείο 19, όχι, δεν είναι το σημείο 19, διορθώνει η πρόεδρος. το βρήκα, το 16, είναι σημείο 16. Εδώ δίνω το λόγο στην Δύο την εισηγήτριά μας, για να μας ενημερώσει σχετικά με τον τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα χτες στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για τη βελτίωση της δυνατότητα μεταφοράς των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, όσοι δεν έχουν δουλειά πια στην αίθουσα και θέλουν να κάνουν πηγαδάκια, εκτός αιθούσης παρακαλώ. Ησυχία. Παρακαλώ, η συγκίτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρέπει να θυμηθώ. Ο Φρεντερίκ Ταρντέν, η Τζιν Λάμπερτς ήταν επίσης και ο Φρεντερίκ στη τεχνική ενημέρωση τουλάχιστον, οπότε βασίζομαι και στη δικιά του τη μνήμη. Καλό είναι που υπήρχε αυτή η στήριξη. Λοιπόν, τι διαπίστωσα. Διαπίστωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαρίστως θέλει να προχωρήσει με αυτήν την ρύθμιση και λίγο πολύ κατάπιε όσα προτείναμε. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, τα περιθώρια είναι πολύ μικρά. Στο Συμβούλιο, το μόνο το οποίο αποφασίστηκε είναι η έγκριση για την διάκριση που γίνεται ε, σε σχέση με τους ξένους εργαζόμενους και τους ε, εργαζόμενους από το κράτος μέλος. Αυτό είναι το γεγονός. Εντάξει, δεν θέλουμε φυσικά να υπάρχει αυτή η διάκριση και ξέρω επίσης στο μεταξύ ότι στο κείμενο έγιναν και αλλαγές από τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Κοιτάξτε, τρία χρόνια μετά. Θέλουμε τη μείωση, εξακολουθούμε να τη θέλουμε και είναι καλό που είναι ανοιχτή αυτή η συνεδρίαση. Κατά πόσο θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε περισσότερο όμως δεν το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. δύο Ήταν το θέμα του ορισμού. Σας το λέω με τα δικά μου λόγια γιατί δεν το έχω μπροστά μου το κείμενο. Τι είναι ένας εργαζόμενος ο οποίος μετακινείται. Είναι κάποιος ο οποίος εργάζεται σε κάποια άλλη χώρα, αλλά υπάρχει και το θέμα της διάρκειας. Πόσα χρόνια. Η Επιτροπή μας λέει είναι καλό για τους εργαζόμενους. Δεν είναι όμως δύο χρόνια, γιατί στα δύο χρόνια πρέπει να φύγει. Στα δύο χρόνια περιορίζεται βέβαια ο εργαζόμενος αλλά έχει να κάνει και με τον ιδιωτικό βίο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος Γάλλος πάει στη Γερμανία και εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό της οδηγίας αυτής, εάν αποχωρήσει, τότε τι δικαιώματα έχει αυτός ο εργαζόμενος για αυτά τα δύο χρόνια που δούλεψε στη Γερμανία. Η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Και κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω και μου υπόθηκε, γιατί θα βοηθήσει αυτό το γερμανικό σύστημα. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο εδώ, το οποίο ίσως μπορούμε να πετύχουμε. αν καλύπτεις τις προϋποθέσεις, όταν ε, σταματήσεις τη δουλειά, τότε μπορεί να επιτρέψει ένα opt-out ο εργοδότης, όταν τελειώσει δηλαδή τα δύο χρόνια, να σου επιτρέψει ένα τρίτο χρόνο. Με τι όμως, εμείς πληρώνουμε πολλά επιδόματα και είναι κάτι στο οποίο με στηρίζουν και οι συνάδελφοι, θέλουμε να υπάρχει ένα ανώτατο όριο, να υπάρχει δηλαδή μία περίοδος που να μην αποτελεί μεγάλο βόρο, όταν βάρος, όταν όμως πρόκειται για μεγαλύτερη περίοδο, τότε προσοχή, μην διαπιστώνουμε ότι αγοράζουν ακριβά αυτοκίνητα όπως έχει συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην την πληρώνουν τα συντοξιδωτικά ταμεία δηλαδή. Αυτά συζητήθηκαν. Ελπίζω ότι το τελευταίο θα διαθετηθεί. Θα δούμε τι θα γίνει με τα άλλα δύο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταρντέν. Σύντομα. Η Ρία καλά συνόψισε τη θέση που είναι κοινή θέση για αυτό το θέμα, να αποφύγουμε τις διακρίσεις. Βέβαια θα είναι δύσκολο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε γνώμη <clears throat> για την τριετή περίοδο. Είναι σημαντικό θέμα, αλλά δεν είδα να υπάρχει άνοιγμα. Υπάρχουν τρία σημαντικά θέματα όπου πιστεύουμε ότι έχουμε περιθώριο να κινηθούμε. Για αυτά τα δύο χρόνια προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Νομίζω ότι εκφεύγουμε του ορισμού. Δεν είναι σωστή αυτή η έννοια των δύο ετών. Και επίσης και κάτι άλλο. Διευκολύνουμε την ε, μεταφορά, καλύτερα να διευκολύνουμε την μεταφορά παρά την ε, αποζημίωση, επιστροφή ας πούμε των ποσών αυτών. Νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία σε μια διαπραγμάτευση. Θέλει κανένα άλλο το λόγο. Όχι. Καλή τύχη για τη συνέχεια της διαπραγμάτευσης στη διαπραγματευτική ομάδα και τώρα τελειώσαμε αυτό το σημείο στη μέση διάταξη και στο σημείο 26 θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης της Γιούτα Steinruck, που είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας για τις ε, πραγματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγή για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη. Στις 18 Σεπτεμβρίου για αυτή την ε, έκθεση ε, οργανώσαμε μία ακρόαση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Η συγγήτρια. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε η πρωτοβουλία της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, να συντάξει μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τις ε, εκθέσεις επιθεωρήσεις εργασίας είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Η παραβίαση έναντι διατάξεων ε, ασφάλειας και υγείας στον χώρο απασχόλησης και όρους απασχόλησης στην Ευρώπη δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Έχουμε στην Ευρώπη όλο και περισσότερες περιπτώσεις για τις οποίες ακούμε και πληροφορούμαστε. Πρέπει άμεσα να δραστηριοποιηθούμε Έχουμε και το άρθρο 9 της, ε, του κανονισμού για την ε, απόσπαση εργαζομένων. Καταδείχτηκε ότι οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι εργασίας είναι το κλειδί για την επιτυχία, για την ε, εκμετάλλευση των εργαζομένων. Και επίσης κλειδί επιβίωσης των επιχειρήσεων που δρούν νόμιμα και εδώ πρέπει να αποκλείεται η κατάχρηση τέτοιων δικαιωμάτων και πρέπει να καταπολεμηθούν. Και υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά από αυτά και συζητάμε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Ισχύει και για τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες απώλειες δισεκατομμυρίων δημοσιονομικά στην Ευρώπη λόγω αυτών των καταχρήσεων. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπήρξαν αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για τον έλεγχο, είτε για τους όρους απασχόλησης, είτε για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας. Και αυτή η έκθεση θέλει να ενισχύσει τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους εργασίας και από την άλλη πλευρά να ενδυναμώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, να, να, καταπολεμηθεί, να καταπολεμηθούν οι στρεβλώσεις, οι καταχρήσεις. Σε πολλές χώρες ε, είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες ελέγχων και επιθεωρήσεων λόγω των περικοπών και πολιτικών λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι είναι όλο και πιο περίπλοκα τα θέματα των συμβάσεων εργασίας, αυτά έχουν όλο αρνητικές επιπτώσεις. Οι κρατικές αρχές δεν μπορούν να ανταποκριθούν πια σε όλα αυτά τα προβλήματα. Σε δύο τμήματα έχω κατανείμει την έκθεσή μου. Πρώτον, αιτήματα προς το εθνικό επίπεδο, προς τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, αιτήματα προς το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υλοποιούν ελάχιστε προδιαγραφέ οι εθνικέ αρχές και στην πραγματικότητα μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς και στην ευρωπαϊκή αγορά πανενοσιακά πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκοί κανόνες και διατάξεις ώστε να καταπολεμηθούν οι αρνητικές εξελίξεις και να μπορέσουμε να έρθουμε στο ύψο των περιστάσεων. Στο εθνικό επίπεδο παριθμούμε αρχέ για αποτελεσματικού ελέγχου. Οι έλεγχοι εργασία να γίνονται από και να μην μην μπορεί κανείς ε, εργαζόμενος το καθεστώς του ή να χάνει το να εξαιρείται από τέτοιου είδους ε, επιθεωρήσεις και ελέγχους. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι πρέπει να έχουν αρκετά στελέχη στη διάθεσή τους. Ε. Πρέπει να μπορούν να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τέτοιες καταχρήσεις. Έχουμε και τα αιτήματα <clears throat> να μπορούν ε, να πληροφορούνται χωρίς έξοδα και δαπάνες για τα δικαιώματά τους ε, και να μπορούν να ε, εισπράττουν τα δικαιώματά τους. Τα κράτη-μέλη πρέπει να προβληματιστούν για τη δημιουργία τραπεζών δεδομένων, όπως θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών από κάτι τέτοιο. Στο Βέλγιο έχουμε θετικά παραδείγματα, τα αναφέρω στην έκθεσή μου. Οι επιθεωρητές εργασίας πρέπει να είναι καλά καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι για προσχηματικές ε, περιπτώσεις που θα αντιμετωπίζουν ε, για τους αποσπόμενους εργαζόμενους πολλές φορές δεν υπάρχει ε, καταχώρηση ή καταγραφή τους κυρίως το φαινόμενο των μη καταγεγραμμένων εργαζόμενων μέσα σε ένα θα λέγαμε παραοικονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει ειδική προετοιμασία να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Έχουμε και συστάσεις προς το ευρωπαϊκό επίπεδο για ευρωπαϊκή δράση. Εισαγωγή μιας υπηρεσίας ε, για διασυνοριακή δίωξη και έλεγχο του, ε, της, για την προστασία των εργαζομένων να καταπολεμηθούν οι εταιρείε που είναι απλά γραμματοκιβώτια και θα λέγαμε επίφαση κάποιας εταιρείας ε, να υπάρξουν διασυνοριακοί έλεγχοι, ώστε να υπάρξουν συζητήσει, Σε όλε τι συζητήσει που έγιναν σε σχέση με τα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. εισαγωγή μια ε, κάρτα ενό δελτίου κοινωνική ασφάλισης. Σε πολλά κράτη έχουμε καλά τέτοια ε, πρώτα μηνύματα. Ένας μηχανισμός έγκαιρη προειδοποίησης, ε, πληροφόρηση για νέε περιπτώσει καταχρήσεων και στρεβλώσεων, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για όλα αυτά και αναφέρουμε επίσης και την εισαγωγή μιας εισαγωγίας ή ε, μιας οδηγίας για τον έλεγχο των ε, εταιριών που δρούν ως διαμεσολαβητές ε, για τη διάθεση εργαζομένων αλλού. Κυρίως καταπολέμηση με κανόνες και διατάξεις του κοινωνικού dumping και ενδεχόμενα κυρώσεις και πρόστιμα άμεσα εις βάρος όσων προβαίνουν σε τέτοιες καταχρήσεις. Κλείσιμο τέτοιων επιχειρήσεων που ζητείται να προχωρεί η Ευρωπαϊκή γιατί όχι και για το κοινωνικό ντάμπινγκ να μην γίνεται το ίδιο, διότι πρόκειται για μια μορφή ε, στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Και εδώ θα μπορούσε από πλευράς ευρωπαϊκών επιθεωρήσεων να υπάρξουν συνοδευτικά μέτρα. Και στην επίσκεψή μας ε, ε, στο εργοτάξιο, γαλλικό εργοτάξιο Λαμονβίλ ακούσαμε τα σχετικά. Είναι μια περίπτωση όπου οι εθνικές αρχές δεν ήταν σε θέση να δουν τι συνέβαινε ακριβώς και να δώσουν συνέχεια στις έρευνες και τα διασυνοριακά θέματα. Αυτό είναι μια σύντομη σύνοψη που έδωσα. Χαίρομαι για τα σχόλια τα οποία θα κάνετε και προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας. Είμαι βέβαια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενδιαφέρον το κοινωνικό ντάμπινγκ να καταπολεμηθεί και προς το συμφέρον των ίδιων των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ε, ε, Κυρία Χάρκιν και μετά Ντανούτα Γιασλοβίνσκα. Ευχαριστώ. Ο συναδελφός μου ζητάει συγγνώμη και θέλει να σας πω δύο λόγια εκ μέρους του. Στο, στους φιλελεύθερους χαιρετίζουμε το γεγονός ότι μπήκαν οι επιθεωρήσεις εργασίας ε, στην ατζέντα. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν πρέπει οι Βρυξέλλες να αναρριθμίζουν αυτό το θέμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα πρέπει βεβαίως να καθοδηγήσουμε τα κράτη-μέλη και τις αρχές επιθεώρησης. Γιατί από την επιτυχία τους εξαρτάται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η κατάσταση στις αγορές των κρατών μελών ε, μπορούν να βελτιωθούν και επομένως θέλουμε τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, προστασία των εργαζομένων όλων των κατηγοριών, ιδίω σε ό,τι αφορά τα πρότυπα εργασία, την καταπολέμηση της, των καταχρήσεων, την πληρωμή την πληρωμή των εισφορών, των μισθών όπως πρέπει κτλ. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμιμες ε, συνθήκες εργασίας ε, και η προστασία σε επίπεδο κράτους μέλους και η διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ισοτιμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εταιρείε και ειδικά οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να επιλέγουν χώρες γιατί ακριβώς έχουν κακές επιδόσεις ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις εργασία και να επιλέγουν να εγκατασταθούν ε, εκεί. Ε, μας ενδιαφέρει λοιπόν αυτή η έκθεση, πιστεύουμε και προσβλέπουμε σε μια έντονη συζήτηση και θα συνεισφέρουμε ε, πολύ επικοδομητικά. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ πρέπει να πω με την εισηγήτρια για τα ότι οι επιθεωρήσεις ε, εργασίας είναι πολύ σημαντικά όργανα. Όταν θέλουμε, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις καταχρήσεις και να προστατέψουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Επίσης ε, θα πρέπει να πάυσουν οι προσχηματικές καταστάσεις και θα πρέπει τέτοιου είδους φαινόμενα όπως για παράδειγμα η παράνομα μειούμενη οι παράνομα μειωμένοι μισθοί να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Εδώ ε, αναφερόμαστε σε παράνομη κατάσταση. Εδώ πρέπει να δούμε τι γίνεται συλλογικά, συνολικά. Δεν πρόκειται για ένα μισθό. Ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μισθοί οι οποίοι θα είναι χαμηλότεροι από τον κατώτατο μέσο μισθό. Επίσης, φαινόμενα κοινωνικού dumping. Αυτή η συζήτηση είναι κάτι που διεξάγουμε ε, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη λοιπόν ότι στην ε, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη οι μισθοί είναι ακόμα πολύ χαμηλότεροι από τους μισθούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ρώτησε η κυρία Στάινμπρουκ πώς είναι δυνατόν με 300 ευρώ να τα βγάζει πέρα ένας εργαζόμενος. Για φανταστείτε ότι σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 300 ευρώ μπορεί να ζει κανείς αρκετά καλά και η έλεγχη είναι πραγματικά αδύρυτη ανάγκη, είναι απαραίτητα στοιχεία. Δεν είναι όμως δυνατόν να είναι ένα μέσο αυτή η έλεγχη ώστε οι αλλοδαποί εργαζόμενοι να προσπαθήσει κανείς να ε, τους ε, ξεφορτωθεί ας το πω έτσι και από την άλλη πλευρά η απόφαση του ΔΕΚ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η νομολογία επιβεβαιώνει ε, μια προσέγγιση σαν αυτήν. Για παράδειγμα έχουμε την κατάσταση που σημειώνεται στη Δανία ε, και στην έκθεση υπάρχουν κάποια στοιχεία με τα οποία δεν συμφωνώ. Για παράδειγμα, το εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τις εργασικές επιθεωρήσεις. Εδώ πάμε πολύ μακριά νομίζω. Ξεπερνάμε τα εισκαμένα. <clears throat> Δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν καμιά δικαιοδοσία και αρμοδιότητα. Όταν επίσης πρόκειται για τους αποσπόμενους εργαζόμενους δεν είμαι καθόλου βέβαια ε, αν, αυτή η έκθεση είναι τόσο, μπορεί τόσο εξειδικευμένα να αναφέρεται στους αποσπόμενους εργαζόμενους. Δεν το πιστεύω αυτό. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι εδώ πάλι ξεπερνάμε τα εσκαμένα αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που προτείνονται που είναι υπερβολικά περίπλοκες θα έλεγα και υπερβολικά δαπανηρές. Επιβαρύνουν υπερβολικά τις ε, διαδικασίες και διεργασίες και την ίδια την ποιότητα των εργασιακών ελέγχων μπορεί αυτό να την πλήξει με αρνητικό τρόπο, να την υπονομεύσει. Θα καταθέσω τροπολογίες ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε αυτή την κατάσταση. Άλλος, κανείς. Και εγώ θα μιλήσω με τη σειρά μου. Να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας, όπου η Επιτροπή μας μπορεί να φωτίσει τη... το θέμα αυτό. Για ένα θέμα, πρόκειται για ένα θέμα που και παλιότερα στην, στα πλαίσια της έκθεσης Tyson ε, μιλήσαμε για τον οδικό χάρτη ε, για την ΟΝΕ και μιλήσαμε για τα διακυβεύματα. Προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά η επιθεώρηση εργασίας. Τώρα διαπραγματευόμαστε κάποια κομμάτια της νομοθεσίας. Είναι μερική αυτή η νομοθεσία, που δεν έχουν σκοπό αυτά τα κομμάτια να καλύψουν το σύνολο των προβλημάτων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Παράλληλα λοιπόν με τις συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, καλό θα είναι να διερευνήσουμε τι θα πρέπει να μπει το κέντρο της εντολής της επόμενης Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Τι θα πρέπει να απασχολήσει όλος ιδιαίτερα την επερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως συμφωνώ με την εισηγήτρια. Η Κομισιόν θέλει να παρέμβει. Δεν εκπροσωπείται η Επιτροπή. Υπάρχει εκπροσώπηση ή όχι της Κομισιόν. Θέλετε να παρέμβετε ή όχι. Η συγγήτρια ξανά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Οι τοποθετήσεις κατέδειξαν ότι η συγγητρια ξανα σας ευχαριστω οι σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν. Ε, θα είναι ενδιαφέροντα τα θέματα, θα δούμε που θα καταλήξουμε. Χαίρομαι ότι υπάρχει συνένεση ότι χρειαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές, χρειαζόμαστε πιο ενισχυμένες διασυνοριακές δραστηριότητες δεν συμμερίζομαι όμως το επιχείρημα ότι οι πρωτοβουλίες είναι υπερβολικά δαπανηρές και υπερβολικά σύνθετες και περίπλοκες. Είδα μελέτες όπου αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές χώρες είναι τριψήφιου εκα, ποσού εκατομμυρίων, διορθώνει η ομιλήτρια, δισεκατομμυρίων. Δηλαδή η απώλεια εσόδων από εισφορές, καταβολές ποσά είναι τεράστια. Δεν είναι εδώ μόνο το θέμα των ελέγχων. Οι, εργα... οι εργασίας πρέπει να καταπολεμήσουν αυτή την κατάχρηση που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στην Ευρώπη και διασυνοριακά στην παροχή υπηρεσιών και παροχή εργασίας από τους εργαζόμενους. Επιτόπου πρέπει να καταπολεμηθεί. Διότι λένε και λέμε ότι είμαστε ανήμποροι αν δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την διασυνοριακή πτυχή στην δίωξη και στους ελέγχους. Και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα καταστήσει πιο διαφανή την όλη υπόθεση. Δεν θέλουμε καταπολέμηση νόμιμων πρακτικών καθόλου. Την παρανομία θέλουμε να πλήξουμε και υπάρχει άμεσα ανάγκη να γίνει αυτό στην Ευρώπη. Έκανα λόγο για τη Γερμανία εχθές. Με 300 ευρώ είπα στη Γερμανία δεν μπορεί να ζει κανείς. Ε, καθόλου, εντάξει, σωστό αυτό. Υπάρχουν και περιπτώσεις από την Ανατολική Ευρώπη. Μια εταιρεία απασχολεί, για παράδειγμα, εργαζόμενους ε, στην Τσεχία για 120 ευρώ κάθε μήνα με τέτοιο μισθό και υπάρχουν πρόστιμα κιόλα όταν δεν βγάζουν πέρα τη δουλειά της βάδιας και αφαιρούν και παρακρατούν ποσά από τον μισθό αυτό των 120 ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα φαινόμενα στις ευρωπαϊκές χώρες. Με την παρανομία αυτή οι εργαζόμενοι βλάπτονται, υπονομεύονται στα δικαιώματα τους αλλά και τα κράτη όσον αφορά εισφορές και ε, ποσά από την κοινωνική ασφάλιση. Πρέπει να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν. Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και η ευρωπαϊκή ενιαία εσωτερική αγορά ανοίγει δυνατότητες για τέτοιου είδους κατάχρηση και παρανομία που πρέπει να καταπολεμηθούν. Ευχαριστώ. Ωραία. Όταν κατατεθούν τροπολογίες θα έχουμε έντονη συζήτηση. Πριν τις 10 Οκτωβρίου πρέπει να κατατεθούν τροπολογίες στις 12 η ώρα. Με ψηφιακή υπογραφή. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 5 Νοεμβρίου τις συμβαστικές τροπολογίε στις 25 και θα ψηφίσουμε την επαύριον. Στις 26 Νοεμβρίου. Τελειώσαμε με το σημείο 26 και πάμε στο σημείο 27. Ξαναδίνω το λόγο στη Γιούτα Στάινρουκ. Θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ έκθεση πρωτοβουλίας πάλι για μια ολοκληρωμένη αγορά παράδοση θεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση της Επιτροπής Ενιαίας ε, Εσωτερικής Αγοράς επικεντρώνεται στην βελτίωση όσον αφορά τα θέματα των καταναλωτών. Η δική μας γνωμοδότηση έχει νόημα και είναι σκόπιμη ώστε τα θέματα των εργαζομένων, γυναικών και ανδρών σε αυτόν τον τομέα να καλυφθούν όπως πρέπει. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια αυξανόμενη αγορά και η διασυνοριακή παράδοση για πελάτες πρέπει να πλουστευτεί. Αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζει κανείς με σαφήνεια ότι δεν μπορεί χωρίς δαπάνες ε, δωρεάν να γίνονται τέτοιες παραδόσεις διασυνοριακά. Ακριβώς και όσον αφορά πακέτα και δέματα. Σε αυτόν τον τομέα ήδη σήμερα υπάρχουν τεράστια προβλήματα λόγω υπεργολαβιών. Για παράδειγμα, όσον αφορά εντολές που δίνονται από, την, ε, από μια επιχείρηση προς άλλους, όμως εργασιακά από την μητρική εταιρεία αποσυνδέονται απόλυτα και έτσι εξοικονομούν και κινδύνους και δαπάνες οι μητρικές εταιρείες. Δεν καταβάλουν ούτε επιδόματα ε, διακοπών, ε, ε, μέρημνας, κανένας δεν έχει τέτοιες υποχρεώσεις λοιπόν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι καλύτερη διασυνοριακή κάλυψη με απλούστευση των ετικετών και της επισήμασης συσκευασιών, βελτίωση υπηρεσιών που παρέχονται από τους εθνικούς παρόχους, όμως πρέπει όλα αυτά να γίνουν σε ένα τακτό, τακτικό πλαίσιο ε, και ε, να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Η αρχή του όλο ταχύτερα, όλο καλύτερα και άμεσα από τις επιχειρήσεις θα πρέπει να αφορά στην εφαρμογή της όλες τις επιχειρήσεις. Σε όλες τις επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται οι εργαζόμενοι στις ανάγκες. Αυτό συναρτάται με την ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, με την ε, επιμόρφωση για τα συστήματα τα ηλεκτρονικά, της ε, εξέβρεση, της συντομότερης οδού, να δούμε και τι γίνεται με το χρόνο εργασίας όσον αφορά τη φόρτωση ενός οχήματος, την εκφόρτωση, την, τον ανεφοδιασμό με καύσιμα. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται αποκλειστικά εις βάρος των οδηγών που είναι ε, couriers ή deliverers ε, και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Προσβλέπω στη συζήτηση και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Θέλει κανένας να πάρει το λόγο. Τη συζήτηση. Να παρέμβει στη συζήτηση. Όχι τροπολογίες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Θα τις εξετάσουμε στις 5 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα ψηφίσει στις 5 Δεκεμβρίου και θα ασχοληθεί η Επιτροπή που θα ψηφίσει για το θέμα αυτό στις 16-17 Δεκεμβρίου. Και πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, σημείο 28, δίνω το λόγο τον Τέβι Κάζα, εισηγητή για γνωμοδότηση για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το λιαπτικό εμπόριο προς όφελος όλων των παραγόντων Μπορείτε να μας παρουσιάσετε, κύριε Κάζα, τις 31 τροπολογίες Ευχαριστώ. Οι τροπολογίες που προτείνουν οι συνάδελφοι δίνουν νέα ενέργεια στο λιανικό εμπόριο και ενισχύουν τα ήδη υπάρχοντα μέτρα προκειμένου να ανταμετωπιστεί η ανεργία στα κράτη-μέλη. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων στους συναδέρφους όλων των πολιτικών ομάδων για τις τροπολογίες τους στο σχέδιο γνωμοδότησης. Σε αυτά θα αναφερθώ και τώρα. Όσον αφορά πρώτον την αναγκαιότητα να λάβουμε υπόψη μας την κινητικότητα στην εργασία και τα ωφέλη για το χοντρικό και το λιονικό τομέα. Επίσης, η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που ζητάει η αγορά και στα προσόντα που έχουν εργαζόμενοι, που είναι η τροπολογία 10. Η έμφαση επίσης που δίνεται στην ευθύνη των εργοδοτών να προετοιμάζουν τους εργαζομένους για κάθε αναδιάρθρωση του τομέα εξαιτία της καινοτομίας. Συμφωνώ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να το ξέρουν από πριν. Επίσης αναφέρεται και η σημασία της διαβίου κατάρτισης. Πολύ σημαντικό σημείο και αυτό. Αναφέρεται σε κάποια από τις Και πρέπει να υπάρξει στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορα μικρά χωριά για τους ηλικιωμένους είναι κάτι που αναφέρεται στην τροπολογία 31. Είμαι επίσης υπέρ πολλών στοιχείων που προτείνει ο Ανδρέα Κοτσολίνο, συναδελφός μου. Τα στοιχεία αυτά διαγράφουν μια πολύ καλή εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η διατύπωση. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά μεταξύ μας για να καταφέρουμε να πετύχουμε την τέλεια διατύπωση. Θέλω επίσης να ευχαριστώ και τον συνάδελφο Καμπαρνό για τις τροπολογίες 3, 16, 20 και 28 και 29. Είναι εξαιρετικές πραγματικά οι τροπολογίες αυτές. Θέλω να ενημερώσω και την Προεδρία και τους συνεδέρφους για το ότι προς το παρόν υπάρχουν τέσσερις συμβαστικές τροπολογίες ήδη, οι οποίες μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει. Συμπεριλαμβάνουν 1, 2, 6, 7, 8 και 9, 16, 17, 18 και 19. Όλες αυτές οι τροπολογίες καλύπτονται από τις συμβατικές. Οπότε, με ενθουσιασμό και αισιοδοξία προσβλέπω σε συνεργασία με τους κοιόδες εισηγητές και τους υπόλοιπους βουλευτές. Και αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη γνωμοδότηση αυτή. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας μέχρι τώρα για όσα μου έχετε πει τις τελευταίες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ποιος θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ, η κυρία Κοστέλο. Μετά, η κυρία Λάμπερτ, όχι. Ωραία, η κυρία Κοστέλο μόνο. Παρακαλώ, κυρία Κοστέλο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η τοποθέτηση είναι από πλευρά σχεδόση Συγητού της των Σοσιαλδημοκρατών κ. Κωσολίνου. Πρώτα απ' όλα μας ζήτησε να διαβιβάσουμε την άποψή του για την έκθεση. Θεωρεί λέει ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Κάζα είναι ένα εξαιρετικό κείμενο. Παρότι λείπουν κάποιες κοινωνικές πτυχές, ε, όλες οι τροπολογίες ε, όμως ε, που έχουν κατατεθεί συμπληρώνουν αυτές, αυτά τα κενά. Ο κύριος Κασολίνο εργάστηκε με τον κύριο Κάζα για συμβαστικές τροπολογίες και έχει την βεβαιότητα ότι θα είναι θετικό το αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον κύριο Κασολίνο είναι πολύ σημαντικές για την ομάδα μας. Πρώτα η τροπολογία 5 που ασκεί στη συμπεριφορά πολυεθνικών εταιριών. Λόγω της οικονομικής ύφεσης υπήρξε σημαντική απώλεια θέσεων απασχόλησης ε, στο λιανικό εμπόριο και ε, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πιέζονται οι εργαζόμενοι να εργάζονται με πιο μικρά ωράρια στην απασχόλησή τους. Και επίσης πρέπει να δούμε ότι εδώ γίνεται χρήση κάποιων συστημάτων ε, επιδότηση όσον αφορά την κάλυψη αυτών των αναγκών. Όσον αφορά τον ελληνικό τομέα που χαρακτηριζόταν με ε, ελαστικότητα και την χρήση ε, προσωρινής εργασίας ακόμα και για την κάλυψη κανονικών εργασιακών αναγκών ακόμα και χρησιμοποιώντας τους εργαζόμενους κατά, τη, κατά και εκτός ωραρίου εργασίας πράγμα το οποίο τους πιέζει ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την κάλυψη των αναγκών όσον αφορά το άνοιγμα ε, καταστημάτων ε, για παράδειγμα κατά τις ε, Κυριακές πρέπει να προστατευτεί το μέσα αυτό. και τα συνδικάτα και η Eurocommerce υποστηρίζει την, προστασία, την παροχή αυτής της προστασίας. Στην τροπολογία με προφορική τροποποίηση μπορέσαμε να διαγράψουμε την τελευταία προ, πρόταση που λέει να μπορέσουν να διασφαλιστούν όροι κανονικού ανταγωνισμού, θεμητού ανταγωνισμού. Και αν υπάρξει αυτή η συμφωνία μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις άλλες ε, τροπολογίες και θέλουμε να τονίσουμε τρεις στόχους. Ε, πρώτον, ε, να αντιμετωπιστούν οι να αντιμετωπιστεί η εξαφάνιση των μικρών καταστημάτων από συνοικίες και από τα κέντρα αστικών κέντρων και να καταπολεμηθεί η επικέντρωση σε μεγάλα καταστήματα. Μετά να δούμε την καταπολέμηση των ατυχημάτων όσον αφορά τον λιανικό τομέα που είναι ένας τομέας που πλήττεται περισσότερο από αυτό το φαινόμενο και ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην οδηγία για την αντιμετώπιση των μειοσκελετικών ε, ασθενειών. Επίσης πρέπει ο τομέας λιανικού εμπορίου να τύχει αύξηση εργασιακών επιθεωρήσεων για να μπορέσει να προστατευτεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς? Όχι. Ο εισηγητής μήπως θέλει να απαντήσει στην κυρία Κοστέλο. Ναι, σύντομα πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σε αυτά τα οποία αναφέρονται από πλευράς του συναδέλφου Κασολίνο για την τροπολογία 5 και την τροπολογία 14, μην αποδεκτά τα σχόλια η τοποθέτηση αυτή. Όπως έχει όμως τώρα η πρόταση, όπως έχει διατυπωθεί, πρέπει να αποσαφινιστεί το πλαίσιό της. Συμφωνώ ότι υπάρχουν σημαντικές τροπολογίες, όμως το κείμενο πρέπει να διευκρινιστεί οπωσδήποτε. Πρέπει να εργαστούμε και να συνεργαστούμε κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη το θέμα της τροπολογίας 14. Επίσης συμφωνώ όσον αφορά την αναφορά που έγινε για τα μικρά καταστήματα και μαγαζιά στα κέντρα χωριών, στα αστικά κέντρα και συμφωνώ ότι μπορώ να μπορώ να δεχτώ αυτές τις τροπολογίες για αυτά τα μικροκαταστήματα σε σχέση με τα μεγάλα. Όσον αφορά <clears throat> για το άλλο θέμα, πρόεδρε, συνάδελφοι, θα συνεχίσω να εργάζομαι για την συμβαστική τροπολογία και ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια λύση που θα υιοθετήσουμε. Ευχαριστώ. Merci Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στις 17 Οκτωβρίου. Θα τις ψηφίσουμε την ίδια μέρα, ώστε να λυθούν υπόψη από την Επιτροπή ΙΜΚΟ, 5 Νοεμβρίου. Δεν έχω τίποτα στα διάφορα. Συνεπώς, θα συναντηθούμε και πάλι στις 10 Οκτωβρίου, 9 με 11.30 στο Στρασβούργο. Είναι 5η πρωί αυτή είναι η επόμενη συνεδρίασή μας και μετά 17 Οκτωβρίου 9 με 12.30 εδώ στις Βρυξέλλες. Καλό σας απόγευμα.